σε όλους τους συναδέλφους. Και τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Στην ε, σημερινή, ε, στην τωρινή φάση έχω μόνο μία αλλαγή να προτείνω. Για την ημερήσια διάταξη ζητά το λόγο. Κοιτάξτε, να ολοκληρώσουμε τα, τις ημερήσιες διάταξης και θα σας δώσω το λόγο. Στην ημερήσια διάταξη για την πέμπτη οι ομάδες συμφώνησαν ο τίτλος του δεύτερου σύστημα, το δεύτερο θέμα για θέματα που αφορούν τις, θα πρέπει να είναι που αφορούν τη Ζιμπάμπουε και τους ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπινών δικαιωμάτων θα είναι το δεύτερο θέμα. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή που προβλέπετε. Δεν ξέρω αν έχετε σχόλια, αντιρρήσεις. Όχι λοιπόν, αποφασίζεται ομόφωνα η ημερήσια διάταξη. Η κυρία Αλφάνο, διαδικαστικό. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω εσά και την ομάδα μου, την Άλντε, γιατί στι 8 Ιανουαρίου, μάλλον πιο συγκεκριμένα στι 7 Ιανουαρίου, το κοινοβούλιο μα χάρη στη δική σα ευαισθησία, επέτρεψε την διοργάνωση μιας επαιτίου της 20 ετίας της ε, δολοφονίας του πατέρα μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συμμετείχαν ε, στο διήμερο αυτό εορτασμό και χάρη στην Άλδη μπορέσαμε να διοργανώσουμε μια διεθνή διάσκεψη των αρχηγών αστυνομία όπου συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του FBI, της 10 και όλων των Ιταλικών αρχών. Ήταν μια διάσκεψη που είχε μέγα αντίκτυπο στον τύπο και θα φροντίσω ώστε να στείλω ψηφιακά στους συναδέλφους ε, το, ένα ανακοινωθέν τύπου για να γνωρίζουν ακριβώς τι συνέβη. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο, εσάς προσωπικά Πρόεδρε και την ομάδα μου, την Άλντε. Σας ευχαριστώ κύριε Αλφανό. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση για τη γεωργία στις άκρος απόκεντρες περιφέρειες. Καταρχάς, έκθεση Παπαστάμκο. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριε